Okay, colleagues, meeting now on... Συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας με το σημείο 22. Αντιπροσωπεία ad hoc στο φόρουμ στις 16 με 18 Ιουλίου. Εγώ, Χωσέ Φαρία, η Τερέσα Χιμένεθ, ο κύριος Σόφκα, η Άνια, η Μιρέγιο, ήμασταν τα μέλη της αντιπροσωπείας. Το φόρουμ υψηλού επίπεδου είναι ο χώρος όπου τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ αναθεωρούν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και κάποιες χώρες παρουσιάζουν τα εθνικά του σχέδια. Η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ισπανία φέτος παρουσίασαν τα, ε, ε, τις εθελούσιες εθνικές εκθέσεις τους. Θα πρέπει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δουν η χώρα τους ε, ποια έκθεση παρουσίασε και τι είπε στα Ηνωμένα Έθνη για του αναπτυξιακού στόχου τη χιλιατίας. Εμείς είχαμε εξαιρετικέ συνεδριάσεις, συναντηθήκαμε με τον κύριο Γκουτιέρε, τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και με τον κύριο Μοταχάμε, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και με τη Λουί Χάρμπορ, η οποία είναι το πρόσωπο κλειδί για τη δράση του ΟΗΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Συναντήσαμε και τον Αχίμ Στάινερ, τον UNDP Administrator Έχετε αντίγραφο της έκθεσης στο φάκελό σας. Το βασικό που πρέπει προφορικά να πω είναι το εξή. Αν συγκρίνω την κατάσταση με το 2015 όπου είχαμε ισοδοξία για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας τους οποίους προσυπέραφε σύσσωμη διεθνή ε, κοινότητα, το θλιβερό φέτος ήταν ότι μέρος αυτής της ε, αισιοδοξία είχε εξατμιστεί γιατί οι ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί από την ε, πολυμερή άγουσα. Και αυτό επηρεάζει τα μάλλα των Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Από ό,τι βλέπω, η εκπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη ε, παρετήθηκε. Σήμερα το απόγευμα έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η τελική διακήρυξη για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας δεν υιοθετήθηκε ομοφόνος, ε, δεν την προσυπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και αυτό είναι δυστυχές, γιατί μπορεί να περάσει η μπάλα, να δοθεί πάσα και σε άλλες χώρες. Και αυτό θα ήταν εξαιρετικά απογοητευτικό. Από εκεί και πέρα, ο Αντώνιο Γκουτιέρας μας μίλησε για τη θεμελιώδη μεταρρύθμιση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυσή του και υπονομεύεται όλη αυτή η προσπάθεια με αυτές τις εξελίξεις. Το κριτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου με δεδομένο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε απομακρύνονται από την πολυμερή προσέγγιση και με δεδομένο ότι επικρατούν εντάσεις αλλού στον κόσμο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις προσπάθειές της να καταλάβει ακόμα περισσότερο χώρο στο θέμα των αναπτυξιακών στόχων τη χιλιετία και των βιώσιμων ως συνέχεια ε, και στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε και την έκθεση IPCC για την κλιματική αλλαγή και πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να προστατεύσουμε τον πλανήτη από την υπερθέρμανση. Επομένως, η διάσκεψη αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί και του χρόνου, το 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει έκθεση για τη συνολική της επίδοση, όχι μόνο αναχώρα, η κάθε χώρα ξεχωριστά. Και από τη στιγμή που τα ηγετικά ενία θα πρέπει να τα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα, ε, πώς θα λειτουργήσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι σε αυτή την πρόοδο. Στη συνεδρίαση των συντονιστών συζητήσαμε αυτό το θέμα. Φέτος, για πρώτη φορά, Έχουμε μια κοινή αντιπροσωπεία στην Νέα με μέλη από τη δική μας Επιτροπή για την Αναπτυξιακή Βοηθεία, με μέλη από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, μεικτή λοιπόν αντιπροσωπεία από δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη όμως καλύπτουν πολλά και διαφορετικά πεδία. Έχουμε HLPF, έχουμε το, την COP, τη διάσκεψη των μερών για την κλιματική αλλαγή και εκεί γίνεται αιτήσια ε, συζήτηση, διάλογος για τους ε, ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους και επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτός ε, θα είναι ίσως ο πρόεδρος ή ο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξού και έχουμε ψήφισμα κάθε χρόνο για το HLPF, για το High Level δηλαδή Forum. Και πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να καταλάβει το χώρο που έχουν αφήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, ο χρόνος πιέζει λοιπόν να δώσω ενδεχομένω το λόγο στους συναδέλφου. Ο Άρνη Ελίζη ήταν εκεί. Είναι μαζί μας. Α, βλέπω και την Άνια. Έχουμε δύο συναδέλφους. Ποιο, ποιος από εσάς θέλει να πάρει το λόγο. Η Άνια ίσως. Δεν μπορείτε ε, να είστε εξαιρετικά ευγενικοί και να παραχωρείτε ο ένας το λόγο στον άλλον και να μην μιλάει κανείς. Άνια, εσύ πρώτη, παρακαλώ. Ή μάλλον ε, ε, εσύ και η Άνια μετά. Ευχαριστώ. Δεν έχω προετοιμάσει ομιλία για το θέμα αυτό. Αυτά που είπατε όμως είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει κάθε χρόνο να είμαστε προετοιμασμένοι και να συντάζουμε έκθεση για το θέμα αυτό. Χάρηκα που πήγα στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε την περασμένη εβδομάδα τα Ηνωμένα Έθνη δημοσίευσαν μία έκθεση η οποία με προβλημάτισε ως προς κάποια σημεία της. Ένα σημείο το οποίο εγώ προσλαμβάνω και αντιλαμβάνομαι ως ένα από τα πιο επίγοντα είναι η παραγωγή και κατανάλωση κρέατος. Σε ό,τι με αφορά εμένα προσωπικά λοιπόν, προσωπική μου αποστολή στη Νέα Υόρκη ε, μπορώ να πω ότι επιτεύχθηκε αλλά ήταν εξαιρετικά σημαντικό που ούτω ή άλλω ήμασταν όλοι εκεί ω μέλη τη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπούσαμε επισήμω και καταφέραμε να ακουστεί ε, στεναρή η αλλω ημασταν ολοι εκει ως μελη τη αντιπροσωπειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ. Ο Άρνη, παρακαλώ. Να τονίσω το οποιο εκπροσωπουσαμε επισήμω και καταφεραμε να ακουστει ε στεναρη η φωνη του ευρωπαικου κοινοβουλιου στη νεα υορκη ευχαριστω ο αρνη παρακαλω να τονισω το εξη κι εγώ. Μιλήσαμε για την κατάσταση των ζώων παγκοσμίω, πώ η κτηνοτροφία ε, χρησιμοποιεί πολλούς πόρου και βλάπτει το περιβάλλον κλπ. Αυτό που κάναμε και άλλοι συναδελφοί όπως ο Γκίντερ, πέρσι η Υόρκη προσπαθήσαμε πηγαίνοντας στην Νέα Υόρκη πολλές φορές να δράσουμε. Και ευχαριστώ την αντιπροσωπεία μας στη Νέα Υόρκη για όλες τις προσπάθειες τους και κυρίως επειδή μας καθοδήγησαν. Χαίρομαι που θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε τον κύριο Γκουτέρες να το δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Γκουτέρε για 10 λεπτά στην ουσία αρχικά, αλλά τελικά ήταν 25 και βάλε. Μιλήσαμε λοιπόν για πολλά θέματα. Μιλήσαμε για την εκθεσή μας για την κλιματική διπλωματία και ο ίδιος ενστενίστηκε αυτό το θέμα και συζητήσαμε πραγματικά θέματα που αφορούν την κοινοτροφία, παραγωγή κρέατος, περιβάλλον, κλίμα. και είδαμε ότι οι ΙΠΑ είχαν αρνητική στάση. Θα θέλαμε λοιπόν εμείς να δράσουμε επειδή εμείς οι ίδιοι πρέπει να δημιουργήσουμε υποστήριξη. Είχαμε και άλλες εκδηλώσεις. Ίδρυμα Μπέτσελσμαν για νέα πρότυπα και νέους μηχανισμούς συλλογής δεδομένων. Και όπως είπε και η Λίντα, οι δύο χώρες που είναι αντίθετες στα αποτελέσματα αυτά είναι το Ισραήλ και η ΕΠΑ. Κάτι το οποίο δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι άλλο που μου φάνηκε θετικό είναι ότι θα έχουμε κοινέ αντιπροσωπίες. Αυτό είναι καλό. Αλλά όπως είδαμε στην έκθεση για την κλιματική διπλωματία δεν υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή. Θα θέλαμε λοιπόν στην Επιτροπή περιβάλλοντο η ΕΦΕΤ να συμμετάσχει με διάσκεψη στο Κατοβίτσε. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε κοινέ αντιπροσωπίες, ιδιαίτερα για τα θέματα του περιβάλλοντος. Να μην έχουμε μόνο μία-δύο επιτροπές, αλλά πέντε-έξι που να εκπροσωπούνται με σημαντικούς εκπροσώπους, γνώστες των θεμάτων, ώστε να φαινόμαστε. Γιατί αυτά τα θέματα πήγαν πέραν του περιβάλλοντος και σε επιτροπής περιβάλλοντος ώστε να μπλέξουμε και άλλους συναδέλφους. Είδαμε από κάποιους συναδέλφους από τη Σουραστική ομάδα κάποιες εκκλήσεις για μια προοδευτική κοινωνία. Αλλά πρέπει όλα αυτά που κάνουμε στο Κοινοβούλιο να φαίνονται, να είναι ορατά το τι συζητάμε, το τι ψηφίζουμε Είπαμε ότι όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Και όπως είπε και η Λίντα, έχουμε και την επόμενη χρονιά μπροστά μας, πολύ σημαντική, γιατί ακόμα η Κομισιόν έχει φτιάξει ένα δικό χάρτη. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι τέτοιο ακόμα από την Κομισιόν και θα πρέπει την επόμενη φορά, το καλοκαίρι, με το νεοκλεγέν Κοινοβούλιο πριν τη νέα Κομισιόν να κάνουμε κάτι. Δύσκολο αυτό βέβαια, αλλά στο σημειώσουμε ότι πρέπει δηλαδή να καλέσουμε την Κομισιόν να δώσει μια καθοδήγηση εκπροσώπησης ώστε να ξέρουμε ακριβώς πώς θα εκπροσωπείται η Ένωση. Να το έχουμε λοιπόν και αυτό υπόψη μας για τις επόμενες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ. Okay, thanks very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιο άλλο. Χέιντι, που ήσουν πολύ ενεργή αυτό το θέμα, παρακαλώ. Λίντα, ευχαριστώ. Θυμάμαι στο Στρασβούργο, στο διάδρομο. Πρέπει να ήταν Νοέμβρη, Δεκέμβρη φέτο, πέρσι μάλλον, είχε σκοτάδι. Και είπες ότι έπρεπε να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης Τώρα, για τους συντονιστές της ΔΕΒΕ και της ΕΜΒΗ, αυτό που έχουμε προετοιμάσει είναι θαυμάσιο. Πολλοί συνέβαλαν σε αυτό και οι επικεφαλής των γραμματιών αυτών των δύο επιτροπών και να τη δουλειά τους. Είμαι βέβαιο λοιπόν ότι αυτή η έκθεση που έχουμε εδώ ότι θα δεχτεί την ισχυρή στήριξη των θεσμικών οργάνων. Αυτό που κάναμε βεβαίως δεν είναι τόσο συστηματικό, παρόλο που ήταν αρκετά ευρηματικό. Πάντως, τώρα ο Πρόεδρος πρέπει να λάβει αυτή την πρόταση και να την αποδεχτεί, να δεσμευτεί. Γιατί πρέπει να συμμετάσχει και αυτό το θεσμικό όργανο στην εφαρμογή. Θα υποστηριχτεί λοιπόν από του συντονιστέ Envy και θα τη λάβει την πρόταση αυτή ο πρόεδρο και μετά θα μπορούσαμε να την παρουσιάσουμε και σε άλλου. Ίσως και εθνικά κοινοβούλια μπορεί να ενδιαφέρονται τα πιο προχωρημένα. Αλλά μπορούμε να τους τη στείλουμε και ελπίζω να έχουμε μια ευκαιρία μετά τις εκλογές, αν θα είμαστε εδώ, να το συζητήσουμε και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τελευταίο, την Πέμπτη, την Πέμπτη έχουμε την πλατφόρμα με την μεγάλη συμμετοχή και το αντίστοιχο έγγραφο προσκέψη εμείς μαζί με την ΕΜΒΗ μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά τέλος πάντων ξαναλέω, είναι εντυπωσιακή αυτή η πρόταση που έχουμε εδώ μπροστά μας. Ναι, για αυτό το φόρουμ με τους πολλούς φορείς Το θέμα είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου. Οπότε ίσως πρέπει να το ερευνήσουμε και να επανέλθουμε μετά την συνάντηση του φόρουμ την Πέμπτη. Επίσης έχουμε το έγγραφο Timmermans και την έκθεση που προβλέπεται για την ανάπτυξη. Οπότε μέχρι τη νέα Κομισιόν πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα γίνει με την Κομισιόν. Θα δημοσιεύσουμε τα έγγραφα που προετοιμάσαμε το 19 πριν σε ευρωεκλογέ. Να μας το πει αυτό η Κομισιόν, αν θέλουν να το σχολιάσουν. Γιατί έχουμε και την ΤΕΦΚΟ κλπ. Αλλά να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε άλλα δύο θέματα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καραβιώνα από την ΤΕΦΚΟ στην μονάδα που παρακολουθεί τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ήμουνα και στην Αγιόρκη, αλλά και στην συνεδρίαση την ενημερωτική που κάνατε τον Ιούλη και στη συνάντηση με τον Επίτροπο Βέλα κατά τη διάρκεια της ε, υψηλού επίπεδου εβδομάδος. Σα ευχαριστώ λοιπόν που υποβάλλατε αυτή την έκθεση και με εντυπωσίασε ο αριθμός, υψηλό αριθμού συναντήσεων που είχατε. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης ήταν πολύ ικανοποιημένη με την αποστολή αυτή και νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ισχυρή δέσμευση του Κοινοβουλίου. Όπως λέτε και εσείς, σε καιρούς που παρουσιάζουν προκλήσεις και επειδή ο ενθουσιασμός υποχωρεί όπως επιστώσαμε ήταν κέριο. Επίσης βέβαια αυτό αντανακλά και τη δέσμευσή μας για παραμονή στην πρωτοπορία της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως είπατε κι εσείς, φέτος και του χρόνου κατά την προετοιμασία βέβαια του φόρουμ του 19. Εμείς από την ΔΕΦΚΟ εργαζόμαστε πάνω σε αυτή την έκθεση. Ήδη έχουμε λάβει κάποιες συμβολές που εξετάζουμε και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και άλλες συνεδριάσεις όπως ξέρετε με κάποια μέλη, Τετάρτη νομίζω, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες από αυτού. Και αυτό το έγγραφο σκέψη επίσης γίνεται κάποια δουλειά. Έχουμε και τα, βραβεία, ευρωπαϊκής, τα ευρωπαϊκά βραβεία βιωσιμότητας, που και αυτό είναι άλλη μια παράλληλη διαδικασία. Όλα αυτά λοιπόν έχουν τεράστια σημασία ενώπιση αυτό, που θα γίνει το 19. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. και εγώ σύντομα να συμπληρώσω από το HSPF. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Κοινοβούλιο για αυτά που κάνει για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Μετά να πω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ σημαντική. Δυστυχώς η υπουργική διακήρυξη έχει παγώσει και η συνένεση που είχαμε με το θεματολόγιο 2030 δεν υπάρχει πια, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και τέλος, να πω ότι ο Νίκ Χέλη ε, πριν από 20 λεπτά ο πρέσβης των ΙΠΑ στο ΝΟΙΕ παραιτήθηκε. Απλώς να σας πω, συνάδελφοι, βλέπετε ότι θα ξανασυναντηθούμε με την Επιτροπή ΕΝΒΗ για να παρουσιάσουμε την αναφορά της παρακολουθησής μας τον Νοέμβριο αλλά και την έκθεση με τις σκέψεις μας. Το πολιτικό κομμάτι Συγγνώμη. Θα υπάρξει δυνατότητα μέχρι την επόμενη συνάντηση του υψηλού πάνελ ε, το νέο κοινοβούλιο να στείλει μια αποστολή. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Πιστεύω ότι στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών θα συμφωνήσουμε, θα υπάρχει συνένεση. Δεν θα είμαι εδώ στην επόμενη Ευρωβουλή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλοι εσείς θα συνεχίσετε να, να διατηρείτε τις προτεραιότητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και να ευχαριστήσουμε και όλους όσους το προσωπικό που βοήθησε ε, σε αυτές τις συνεδριάσεις. Περνάμε στο σημείο 23 και οι δύο ερωτήσεις προέρχονται από μένα, επομένως μπορώ να είμαι και πάρα πολύ γρήγορη. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τα παιδιά πρόσφυγες από την ε, Συρία Απλά να πω ότι δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην Επιτροπή μας στην ανάγκη για εκπαίδευση. Αυτό έχει να κάνει με την δέσμευση που έχουμε αναλάβει να στηρίξουμε οικονομικά την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων από τη Συρία. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν τι γίνεται με αυτά τα χρήματα που έχουν, ε, είχαν δεσμευτεί ότι θα δώσουν. Τι, τι συμβαίνει, γιατί πόσα μιλάμε. Ε, δεν έχω ονόματα ε, για τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Είναι ο Μάικλ Μίλλερ που παίρνει το λόγο από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνατε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη δεύτερη συνεδρίαση των Βρυξελών, τον Απρίλιο που μας πέρασε, σε συνδυασμό με τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί ήδη για το 2018 προστέθηκαν και 21,2 δισεκατομμύρια δολάρια με τη μορφή δανείων από διάφορους διεθνείς εταίρους, χρήματα που πηγαίνουν στην Αίγυπτο, στο Ιράκ και στο Λίβανο. Οι περισσότεροι δωρητές οι στόχοι μπορούμε, να τους γνωρίζουμε εφόσον γίνουν οι δωρεές. Η Επιτροπή από το 2017 έχει αναλάβει να εντοπίσει όλες αυτές τις δωρεές. Αυτό είναι ένα εργαλείο για μας για να μπορούμε να παραμένουμε ενήμεροι, αλλά να ενημερώνουμε και τις χώρες για όλες αυτές τις χορηγίες εκ μέρου των δωρητών. Από τον προηγούμενο Απρίλιο έχουμε εκθέσει τρεις τέτοιου τύπου αναφορές. Η τελευταία δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο πριν την ε, Σύνοδο Κορυφής των, της Γενικής Γραμματείας. 4 δισεκατομμύρια ευρώ εντοπίστηκαν το μεγαλύτερο κομμάτι των δωρεών αυτών κατευθύνθηκε προς διάφορες δραστηριότητες και το 15% των συνολικών δωρεών κατευθύνθηκε προς την εκπαίδευση. Μετά έχουμε την υποδομή, το φαγητό 15%, 14% με συγχωρείτε περίπου. Όταν αναφερόμαστε στην εκπαίδευση, αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει απολύτως δεσμευμένη να βοηθήσει τα παιδιά πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μεσοπρόθεσμα αυτή τη στιγμή λειτουργούμε και προσπαθούμε να αναπτύξουμε στρατηγικές για, τον, για την αναδόμηση του συστήματος της εκπαίδευσης. Είναι αρκετά σημαντικός ο αριθμός των προσφύγων. Προσπαθούμε επίσης να κινητοποιήσουμε ποσά. Παραμένουμε ευθυγραμμισμένοι με την ε, στρατηγική ε, για την εκπαίδευση σε ε, επίγουσες περιόδους όπως αυτή παρουσιάστηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Μεγάλο κομμάτι των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων σχεδιάζονται από τους ίδιους τους δωρητές σε συνεργασία με τις χώρες όπου βρίσκονται οι πρόσφυγες. Ένα άλλο σημείο που θέλω να θίξω στόχος αυτός του να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι όλα τα παιδιά έχουν ε, πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι πάρα πολύ δύσκολος να επιτευχθεί και ο λόγος είναι ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους Σύριους πρόσφαγες συνδέεται και με τις δυσκολίες καταγραφής, μόνιμης κατοικίας, έλλειψης ε, νόμιμων διαδικασιών για τους γονείς των παιδιών, που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά αυτά καταλήγουν να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης παιδικής εργασίας ένα ιδιαίτερα πολυπλοκό ζήτημα. Είμαστε όμως απολύτως αποφασισμένοι να επιτύχουμε όσα περισσότερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που βρίσκουμε στο δρόμο μας για να εξασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά πρόσφυγες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ε, ποιοτική εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται και στις διαβουλεύσεις συνεργασίας που έχουμε με πάρα πολλές χώρες της ε, Μέσης Ανατολής, με τη ε, Ιορδανία, το Λίβανο και άλλες. Μία ερώτηση λέει η Πρόεδρος. Είπατε ότι το 15% αναλογεί στην εκπαίδευση. Οι εκθέσεις αυτές α, αναφέρουν ποια χώρα δίνει πόσα χρήματα και μπορούμε να δούμε τι ποσοστό της κάθε χώρας πηγαίνει στον κάθε Μπορούμε δηλαδή να πούμε πόσο της εκατό του ποσού που δίνει η Γερμανία αντιστοιχεί στην εκπαίδευση. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι εκθέσεις αυτές δεν υπησέρχονται σε τέτοιου τύπου λεπτομέρειες ή ανάφορες. Έχουμε λεπτομερείς εκθέσεις, γιατί όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, έχουμε πάμπολα στοιχεία τα οποία δεν δημοσιεύουμε. Αν θέλετε να έχετε πιο ακριβείς πληροφορίες, μπορούμε να, τι, να σας τις δώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το 2016, σε μια συνεδρίαση, είχαμε δεσμευτεί ότι όλα τα παιδιά θα βρίσκονται στο σχολείο μέχρι σήμερα παιδιά προσφύγων. Σήμερα όμως 43% των παιδιών αυτών παραμένει εκτός εκπαίδευσης, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει στο στόχο μας και άλλη μια σχολική χρονιά ξεκίνησε. Ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση την Επιτροπή. Ξέρω ότι, κάνετε, ότι έχετε βάλει τα δυνατά σας. Έχουμε άλλη μια ερώτηση για την θυματίωση. Στη Νέα Υόρκη συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της ε, TB Alliance όπου μας είπαν ότι η φυματίωση είναι η πιο α, θανατηφόρα ασθένεια στον κόσμο, σκοτώνει περισσότερους από τη μαλάρια και το AIDS σε άθροισμα. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ από την αρμόδια DG. Ο Γιάν Πέλερ είναι εδώ. Συμφωνούμε, λέει, με την αξιολόγησή σας για την ασθένεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στις πρώτες γραμμές ε, στο μέτωπο του πολέμου αντίον της φυματίωσης και τα κράτη-μέλη συμβάλλουν ε, οικονομικά σε περισσότερο από το 50% των ε, χρημάτων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της φυματίωσης. 475 εκατομμύρια ευρώ το 2017 δεσμεύτηκαν για την καταπολέμηση της φυματίωσης. Η Επιτροπή μας εχθές α, έχει, εχθές πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα 5 εκατομμύρια άτομα που έπασαν από θυματίωση θεραπεύτηκαν. Συνεπώς, το 2019 θα φροντίσουμε να κατευθύνουμε ε, ανάλογα ποσά στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση της Θυματίωσης, όπως έχουμε δεσμευτεί και στην πολιτική μας δήλωση ή φυματίωση μπορεί να επηρεάσει τον καθένα σε οποιοδήποτε σημείο. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε μια σειρά από χώρες για να μπορέσουν να προβλέψουν και να θεραπεύσουν ε, σοβαρές ασθένειες όπως είναι η φυματίωση. Όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα για την ε, καταπολέμηση της φυματίωσης. Μια αρρώστια που πλήττει κυρίως τα φτωχότερα στρώματα και τα πιο περιθωριοποιημένα. Η επένδυση στην έρευνα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική, να έχουμε αποτελεσματικά αλλά και οικονομικά φάρμακα. Επίσης χρειαζόμαστε καινούργια διαγνωστικά εργαλεία στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο περιλαμβάνει επενδύσεις και για καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία και εμβόλια, αλλά και εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την αρρώστια. Τέλος, η Κομισιόν θα προσπαθήσει να στηρίξει την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της θυματίωσης, την αύξηση των οικονομικών μέσων, θα καταστήσει πιο αποτελεσματικό το τρόπο που μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παγκόσμιο Ταμείο Καταπολέμησης της θυματίωσης. Από μαζί με άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, για αυτήν την αναφορά, για την εκθεσή σας. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Να ενδυναμώνουμε τα βασικά συστήματα για την καταπολέμηση τέτοιων ασθενειών είναι πολύ σημαντικό. Περνάμε στο σημείο 24. Δεν υπάρχει τίποτα. Το επόμενο, η επόμενη τακτική μας συνάντηση είναι στις 19 Νοεμβρίου στις 3.30. Η επόμενη έκτακτη συνεδρίαση είναι στο Στρασβούργο στις 12 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Δυστυχώς δεν υπήρχε άλλο κενό γιατί υπάρχουν ψηφοφορίες. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για το Horizon 2020. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί σύσκεψη των συντονιστών. Παρακαλώ φύγετε από την αίθουσα όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.